Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε τώρα. Κριστίνα, παρακαλώ. Κύριε Μόργανο, συγγνώμη γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ησυχία παρακαλώ. Έχετε πάρει θέσεις όλοι. Ωραία. Είναι και Δευτέρα απόγευμα, δεν είναι πολύ εύκολο να έχουμε εδώ όλους τους συναδέλφους, αλλά έχουμε τους πιο διακεκριμένους εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω θερμά, να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς μας προσκεκλησμένους. Όλοι εσείς γνωρίζατε πάρα πολύ καλά τον Ken Loach. Είναι γνωσμένο κύριος καλεσμένος μας. Ε, θα περάσω στα Ιταλικά μετά. Έχουμε τη Σελήν Σιάμα, η οποία συμμετείχε στο Αβραβία Λούξ με την ταινία «Τα κορίτσια». Μια εξαιρετική ταινία, ήταν εφινελίστ ε, το 2013 και έχουμε εδώ και τον Ανδρέα Σέγκρε με το έργο που παρουσίασε στα βραβεία Λούξ, ένα πολύ συγκινητικό έργο, η Σουν Λί και ο ποιητής, ε, και κέρδισε το βραβείο Λούξ ε, το 2012. Και επίσης έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας εδώ την Doris Πακ, η οποία όπως όλοι γνωρίζετε ε, έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, αλλά είναι και είναι και η μητέρα όλων ε, ε, και του βραβείου Λουξ κυρίως ε, και τώρα ε, της έχει αναθέσει ο πρόεδρος Σούλτς να είναι συντονίστρια των βραβείων Λουξ και την ευχαριστώ για την παρουσία της εδώ. Και τώρα θα περάσω στα Ιταλικά. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι, περήφανοι και συγκινημένοι που έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που εκφράζει την ύψιστη ε, ευρωπαϊκή σκηνοθεσία. Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για ένα μεγάλο πρωταγωνιστό του, πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού σινεμά που μας άφησε σήμερα. Αναφέρομαι στον Αντρέι Βάιντα, ο οποίος ε, ε άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στα 90 του χρόνια, ένας μεγάλος πολωνός σκηνοθέτης, ο οποίος ε, με το μοναδικό του στυλ ε, γεμάτο πνευματικότητα, ναι. αλληγορία και προσοχή στις ιστορικές δυνάμεις και της χώρας του, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ε, πραγματικά αποτέλεσε μια ελεύθερη φωνή και μια ίσως και άβολη μαρτυρία του τι ακριβώς ε, συνέβαινε στη χώρα του. Ε, να υπενθυμίσω ότι έλαβε και χρυσό φίνικα το 1976 με τον άνθρωπο από μάρμαρο και μετά το 1981 με τον άνθρωπο από σίδηρο, τον οποίο είχε αφιερώσει στο ήταν το σύμβολο μιας ε, Πολωνίας ε, εξοργισμένης, πάντα πρόσεχε την ιστορία της ε, χώρας του και πάντα κατάφερε να τη διηγηθεί με ένα πολύ πνευματικό και συμβολικό τρόπο και με μεγάλη αυστηρότητα. Ήταν και ε, σεναριογράφος και διευθυντής του Θεάτρου της Βαρσοβίας. Ε, το 2000 πήρε τιμητικό Όσχαρ και ε, ε, Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, επίσης το 2001. Είναι μία ακόμα από τις αναγνωρίσεις που έλαβε και επίσης ε, πρέπει να πω ότι πρέπει να αποτίσουμε και φόρο τιμής στον άνθρωπο αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να το αποτίσουμε φοροτιμή και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτή την εξαιρετική φυσιογνωμία που ήταν και ε, ένθερμος ευρωπαϊστής. Ε, ένα χειροκρότημα τουλάχιστον. Ε, και Μπορεί στη συνέχεια στο ε, Παρλαμεντάριο να δούμε και ένα μικρό βίντεο ε, στη μνήμη του Αντρέι Βάιντερ. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά αγαπητοί προσκεκλημένοι, γιατί γιορτάζουμε τα 10 χρόνια του βραβείου Λουξ, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σκηνοθεσίας, το οποίο θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατάφερε ίσως να προβλέψει και την ανάγκη που διαπιστώνουμε σήμερα για μια πιο πλούσια ευρωπαϊκή ε, κινηματογραφία που να αναφέρεται και στα ο πλούτο της Ευρώπης αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτισμός. Τα τελευταία χρόνια φιλοξένησε 100 ε, δημιουργούς αλλά και 100 διαφορετικά οράματα της σύγχρονης Ευρώπης με μια πρωτότυπη ματιά του ευρωπαϊκού ε, σινεμά. Αποφασίσαμε να το γιορτάσουμε με κάποιους εκ των πρωταγωνιστών. Τον Ken Loach, ο οποίος έχει πάρει δύο φορές ε, χρυσό φίνικα, φέτος με το εγώ Daniel Blake, μια διήγηση κρίση, της φτώχειας και της αξιοπρέπειας. Ε, μια πολύ ανθρώπινη ταινία και ιδιαίτερα κοινωνική. Ε, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ και επίσης... Ε, Όπω είπα προηγουμένω, θα ήθελα να ευχαριστήσω και του άλλου δύο σκηνοθέτε, τον Αντρέα Σέγκρε, τη Ελίνη Σαμά και φυσικά την Τόρι. Είναι δημόσια πραγματικά αυτή η συνεδρίαση, γιατί μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο, αλλά και στο Άρτε Σίνεμα, το οποίο ευχαριστώ για την προσοχή του. Το βραβείο Λουξ ε, είναι ένδειξη της προσοχής που προσδίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον πλούτο του ευρωπαϊκού σινεμά, ε, στη θεματολογία του, στην ευαισθησία και στην ε, δημιουργική γλώσσα. Αλλά επίσης κατάφερε μέσω της διέστησης ε, που ε, είχε να υποτιτλήσει τις ταινίες της 23 επίσημες γλώσσες, όχι μόνο των νικητών, αλλά τα τελευταία χρόνια και των ε, τριών ταινιών που είναι μεταξύ των φιναλίστ. Έτσι προωθεί λοιπόν την πολυγλωσσία που είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν ήταν ευρωπαϊκή μόνο, αλλά ορισμένες φορές ξεπέρασε και τα σύνορα της Ευρώπης. Πολλές ταινίες του έγιναν γνωστές και εκτιμήθηκαν και συζητήθηκαν και σε άλλες χώρες εκτός από τη χώρα καταγωγής τους και μπόρεσαν να πρωταγωνιστήσουν και σε διεθνή φεστιβάλ ε, συλλέγοντας επιτυχίες και εκτός του ευρωπαϊκού χώρου αλλά και πιο γνωστοί σκηνοθέτες συμμετέχαν. Ε, κάποιοι εξ αυτών είναι και εδώ στα Βρατσβία Λούξ και νομίζω ε, και θα μας το πούν και οι ίδιοι ε, κατάφεραν έτσι να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ένα διαφορετικό κοινό και εντός και εκτός Ευρώπης. Να υπενθυμίσω ότι ε, κάποια από τις ταινίε που πήραν βραβείο Λουξ ε, πήραν και βραβείο Όσκαρ. Το Ιντ, ο γιος του Σαούλ ε, και αναγνωρίστηκαν ως εξαιρετικές ταινίε. Τα τελευταία αυτά δέκα χρόνια χάρη και στη δική σας τη συνεργασία ε, δηλαδή και το προσωπικό που είναι παρόν, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα βραβεία Λουξ και πάρα πολλοί ευρωβουλευτέ που δεσμεύτηκαν. Θα θέλαμε περισσότεροι βέβαια να συμμετέχουν, η Ντόρι Πακ και άλλοι. είδαμε το βραβείο Λουξ να κάνει γιγαντιαία άλματα. Οι μέρες ε, βραβείων Λουξ ε, ήταν εξαιρετικές μέρες. Ε, πέρσι είχαμε πάνω από 50 πόλεις οι οποίες μετάδωσαν τις τρει ταινίε που ήταν στην τελική ευθεία με σημαντική συμμετοχή και του Ευρώπα Σίνεμα το οποίο ευχαριστώ και που είναι παρόν σήμερα. Σήμερα λοιπόν ε, θα έχουμε και τους φιναλίστ ε, της ε, φετινής έκδοσης. Πρόκειται για ταινίες οι οποίες είναι συμπαραγωγές με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η ζωή μου ως κολοκυσάκι, το όταν ανοίγω τα μάτια μου και το τι Μέρμαν. Είναι τρεις ταινίες ο νικητής θα επιλεγεί από τους ευρωβουλευτές, όπως γνωρίζετε, χάρη στην ψήφο τους και θα προγραμματιστούν ε, επισήμως, ε, θα μεταδοθούν, ε, θα ανακοινωθεί ο νικητής στο Στρασβούργο. Επίσης, τα βραβεία Λούξ, οι ταινίες Λούξ συμμετέχουν σε σημαντικά φεστιβάλ, αλλά υπάρχει και με συνεργασία με το Κάρλο Βιβάρη και με το Φεστιβάλ της Βενετίας. Είναι η πρέσβης μας λοιπόν στα βραβεία Λούξ και ευχαριστώ και το Ευρώπα Σίνεμα γιατί βρίσκονται ε, και στην κριτική επιτροπή αυτών των σημαντικών εκδηλώσεων. Να ευχαριστήσω και τους πέντε νέους συνεφίλ που είναι εδώ. Σηκωθείτε για να σας δούνε. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί αυτά τα νέα παιδιά είναι αυτά τα οποία προωθούν στην Ευρώπη την ευρωπαϊκή ε, κινηματογραφία. Ε, σήμερα θα είδατε ίσως στην ε, στο προάβλιο του Κοινοβουλίου ε, την παρουσίαση. Ε, σήμερα στις 7 η ώρα θα γενιάσουμε μια εξαιρετική έκθεση για τα βραβεία Λουξ που είναι αφιερωμένη στις 100 ταινίες και στους 100 δημιουργούς που συμμετείχαν στα βραβεία Λουξ και υπάρχει και μια εκδήλωση που καταδεικνύει από μόνη της πόσο σημαντικό είναι το βραβείο Λουξ και πόσο αυξήθηκε. Θα υπάρχει μια πραγματικά ευρωπαϊκή εκδήλωση, η προβολή ταυτόχρονα στις 28 χώρες μέλη ε, σύνδεση λοιπόν την ίδια ώρα της ταινίας Mustang ε, με υπότιτλους φυσικά στις 24 επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, θα υπάρχει σύνδεση με το σινεμά Γκαλερί των Βρυξελών, το Γκαλερί de Bruxelles, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Δείχνει λοιπόν τι δύναμη έχει το σινεμά που μπορεί να παρασύρει πέρα από γεωγραφικούς ορίζοντες και γλωσσικούς ορίζοντες και θέλουμε να υποστηρίξουμε το ανεξάρτητο ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό σινεμά και με τη δέσμευσή μας αυτές τις ημέρες, ώστε να δημιουργηθεί ένας πραγματικός χώρος ε, του ευρωπαϊκού σινεμά, να είναι πιο ισχυρό και να ενισχύσουμε και την πολιτιστική, κινηματογραφική και οπτικοακουστική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βραβείο Λουξ βέβαια ε, βασίζεται κυρίως ε, στο φως, όπως το λέει και η ίδια η λέξη. Λουξ είναι φως στα λατινικά. Δώσαμε σημασία σε κάποια θέματα τα οποία είναι περίπλοκα, και προσφέραμε θέματα προς συζήτηση και συζήτηση και στις πολιτικές των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον της κρίσης της Ευρώπης που είναι μια δεντολογική, ηθική, πολιτισμική και κοινωνική κρίση αλλά και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη Ευρώπη, τη παγκοσμιοποίηση, τη μετανάστευση, τις ανισότητες ε, την ανεργία των νέων, τις ε, νέες και παλιές διακρίσεις, αλλά και πάρα πολλές ελπίδες και πολύ μεγάλη θέληση για μια Ευρώπη που θα ανταποκρίνεται περισσότερο στα όνειρα αυτών που την επινόησαν σε δύσκολους, χαλεπούς καιρούς και πιστεύω ότι το σινεμά μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να ερμηνεύσουμε λίγο ευρύτερα και μας βοηθά να ε, δημιουργήσουμε και κάποιους πιο ενδιαφέροντες ορίζοντες που ίσως σήμερα από μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε μπορούσαμε να διαβλέψουμε. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι το να στοιχηματίσουμε και να επενδύσουμε στο ευρωπαϊκό σινεμά αποτελεί ένα σημαντικό ε, βήμα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την Ευρώπη του σήμερα. Δεν μπορούμε να έχουμε Ευρώπη χωρί το σινεμά τη και θα ολοκληρώσω λέγοντα δύο πράγματα. Πρώτον, χαίρομαι διότι και σε μια Ευρώπη που φαίνεται να χάνεται το κεντρικό στίγμα του πολιτισμού, στην τελευταία ομιλία του για την κατάσταση τη Ένωση, ακούσαμε τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ να λέει ότι οι δημιουργοί μα είναι αυτοί που βρίσκονται ε, στα διαμάντια της κορώνας. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να μπορέσουν να προσφέρουν πολιτισμική ποικιλομορφία στην Ευρώπη αυτή είναι η δημιουργία. Και υπάρχει τουλάχιστον ένα καλό νέο. Ε, την τελευταία χρονιά το Ευρωπαϊκό Σινεμά είχε εξαιρετική απόδοση. 180 εκατομμύρια εισιτήρια απολύθηκαν στις αίθουσες, αλλά πέραν αυτού υπάρχει και αύξηση κατά 8% και το 30% των ευρωπαϊκών ταινιών, των ταινιών αυτών συγγνώμη, είναι ευρωπαϊκές. Ε, μέσω του προγράμματος ε, Mediatic, το οποίο θα γιορτάσουμε ε, τα 20 χρόνια του φέτος, θέλουμε να συνεχίσουμε λοιπόν να υποστηρίζουμε την κυκλοφορία, την παραγωγή και την ε, παιδεία στο σινεμά. Ε, το καθήκον που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα λοιπόν οι σκηνοθέτε και με αυτό ολοκληρώνουν, αλλά σκηνοθέτε με τη δική σα την ευαισθησία, ε, το δικό σα το κύρο, ε, τη δέσμευση και ίσω και το γεγονό ότι παρουσιάζεται κάποια άβολα θέματα, όπω αυτά που παρουσιάζει ο Κεν Λότ, ο οποίο πρωταγωνιστεί σε αυτά τα θέματα, είναι και ηθικό ζήτημα. Πρέπει σήμερα να χτίσουμε γέφυρε, γέφυρε αλληλοκατανόηση, διαλόγου, αμοιβαία αναγνώριση για μια Ευρώπη η οποία αρχίζει να ξαναδιεκδικεί σύνορα, που ε, υψώνει τύχη και ε, την οποία ορισμένες χώρες όπως η δική σας αγαπητέ Ken load θέλουν να εγκαταλείψουν. Ε, χάρηκα ιδιαίτερα διότι και εσείς και αρκετοί άλλοι διανοούμενοι και νέοι και το λέω σαφέστατα ε, συνεχίζουν τη μάχη, αλλά εντός της Ευρώπης. Ε, τα πράγματα φαίνονται διαφορετικά, αλλά ελπίζω ο πολιτισμός και η παιδεία να είναι οι μεγάλοι τομείς ε, πάνω στους οποίους θα μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε και να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο όπου οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα θα γίνονται σεβαστά. Να δώσω τώρα αμέσω το λόγο σε εσά, κύριε Λόουτς. Αναμένουμε με αγωνία την παρέμβασή σας και από εκεί και πέρα να πω ότι θα δώσω τη δυνατότητα στους συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν να απαντήσουν στην παρέμβασή σας και μετά θα δώσω το λόγο στην Τόρις Πακ αν θέλει να παρέμβει και να θέσει και κάποιες ερωτήσεις ε, στους ε, δύο σκηνοθέτες μας, τη Σελήν Σαμά και στον Ανδρέα Σέγκρε για να συνεχίσουμε μια συζήτηση η οποία κατά την άποψή μας θα είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Να σας δώσω το λόγο λοιπόν κύριε Λόουτς. Παρακαλώ. Thank you. And, um... Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το προνόμιο που μου δίνετε να έρθω εδώ και να σας πω δύο λόγια. Να πω ότι με τρομάζει κάπως το πολυπληθές κοινό. Καταρχάς, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έμαθα τα δυσάρεστα νέα για τον Άντρεϊ Βάιντα μέχρι να το ακούσω από εσάς. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τα θερμότατα συλληπιτήριά μου για έναν σπουδαίο σκηνοθέτη, πολύ επιδραστικό και για μένα και για τους φίλους μου και για όλους ε, όσοι αγαπούν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Ήταν ένας από τους μεγάλους σκηνοθέτες και μας δίδαξε πάρα πολλά. Μας έμαθε την ιστορία της Πολωνίας και την ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν ένα υπόδειγμα και ήταν έμπνευση για όλους όσοι εργάζονται στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Ευχαριστώ Αντρέ Βάιντα. Καλή αντάμωση. Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό ο τίτλος βραβείο Lux, Lux, φω στα λατινικά. Το φως είναι πολύ σημαντικό για τον κινηματογράφο. Το Σελιλόντ είναι αυτό που μας ε, δίνει τη δυνατότητα να έχουμε κινηματογράφο. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ο κινηματογράφος πρέπει να ρίχνει φως να ρίχνει φως σε ιστορίες, σε χαρακτήρες, να μας διαφωτίζει, να δίνει τροφή για δημόσια συζήτηση. Είναι λοιπόν ο ρόλος του κινηματογράφου και να δίνει και να παίρνει. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι αξίες του διαφωτισμού βρίσκονται υπό αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε. Και η λογική πάνω από την τυφλή πίστη είναι κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τις αξίες οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για εμάς. Ιδιαίτερα για εμάς εδώ. Και πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ και οι βουλευτές στην πατρίδα μου να είχαν αυτή την άποψη. Δυστυχώς όμως όχι. Το φως όμως μπορεί να είναι ψυχρό, μπορεί να έχει ρόλο απλού παρατηρητή. Για τον κινηματογράφο χρειάζεται όμως ζέστη. Πρέπει να δημιουργήσουμε ζέστη, ζεστασιά για τον άνθρωπό μας, συμπόνια, αλλά πολλές φορές αυτή η θερμότητα μπορεί να είναι και θυμός. Θυμός όταν κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε τι συμβαίνει. Το φως λοιπόν είναι πολλά πράγματα. Και θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για τρία πράγματα. Να μιλήσω καταρχάς λίγο για τον κινηματογράφο και τι μπορεί να κάνει. Και ιδιαίτερα για το τι μπορεί να κάνει ο Βρετανικός κινηματογράφος, τι χρειάζεται από την Ευρώπη, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω και για το δίλημα της αριστεράς, σε ό,τι αφορά το Βρετανικό δημοψήφισμα, γιατί νομίζω πως εδώ έχει γίνει μία παρεξήγηση και δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα αρκετά αμφιλεγόμενο θέμα, να σας ε, πω δηλαδή μερικές ειδήσει από την πατρίδα μου που ίσως να μην έχετε μάθει με τον τρόπο που έγιναν. Ακριβώς γιατί νομίζω πως υπάρχουν κάποια προβλήματα επικοινωνίας με τον τύπο, με τα μέσα ενημέρωσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει, το οποίο μπορεί να διαφέρει από αυτά που έχετε εσείς ακούσει και διαβάσει. Αρχίζουμε λοιπόν με το κινηματογράφο. Ό,τι και αν πει κανεί για τον κινηματογράφο, η αλήθεια είναι ότι είναι το πιο υπέροχο, θαυμαστό μέσο. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς εδώ σήμερα. Μας ε, ενδιαφέρει, πονάμε αυτό το μέσο, γιατί πιστεύω ότι ο κινηματογράφος έχει τα πάντα. Έχει και το δράμα, έχει τους χαρακτήρες, τους ήρωες, έχει τις ιστορίες του, έχει τη λύτρωση, έχει τα προβλήματα, έχει οπτική εικόνα, μπορεί να ενημερώσει, μπορεί να εμπνεύσει τη φαντασία, μπορεί να είναι σουρεαλιστικός, μπορεί να είναι ιστορικός, μπορεί να κάνει τα πάντα, να χρησιμοποιήσει μουσική, να χρησιμοποιήσει κάθε είδος τέχνης, να ενώσει τα πάντα στον κινηματογράφο. Και πιστεύω πως είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι του κόσμου εμείς που μπορούμε να δουλέψουμε στον κινηματογράφο, γιατί είναι μια εξαιρετική μορφή τέχνης που δεν πρέπει να υποτιμάται. Ωστόσο υπάρχουν και προβλήματα και ένα πρόβλημα πιστεύω περισσότερο από όλα είναι το δίλημα που έχει ο κινηματογράφος ανάμεσα στο να είναι ε, εμπορεύσιμο είδος ή να είναι τέχνη. Σε γενικές γραμμές θεωρείται εμπορεύσιμο είδος, θεωρείται μια επένδυση και θεωρείται μάλιστα μια ακριβή επένδυση, ένα ακριβό αγαθό και όσοι επενδύουν στον κινηματογράφο εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια. Κοιτάζουν την παραμικρή λεπτομέρεια έτσι ώστε να αξιολογήσουν την επένδυσή τους. Και ακριβώς ε, γιατί θεωρεί το κινηματογράφος ως επένδυση, διακυβεύεται, τόσο περισσότερο διακυβεύεται η ακεραιότητά του. Γιατί απομακρυνόμαστε πάρα πολύ από την κεντρική ιδέα μιας ταινία. Και όταν γίνεται λόγο για μια ταινία πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίε Και σκεφτείτε, μια ταινία πόσο είναι εμπορικό αγαθό και πόσο είναι μια ιδέα, μια αφήγηση, ένα δράμα, μια τραγωδία, μια κομμωδία. Πώς έχει επηρεαστεί λοιπόν η τέχνη, ένα, μια ταινία, ένα έργο από την ε, ιδιότητά της ως εμπορικό αγαθό. Αυτή τη στιγμή επίσης να πω πως η κουλτούρα της ε, Αμερικής μας έχει, μας έχει πλημμυρίσει και αυτό είναι πρόβλημα. Όπως ίσως γνωρίζετε και από άλλες περιπτώσεις, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θέλουν εταίρους, δεν θέλουν συνεργάτες, αλλά θέλουν υπηκόους, υποτακτικούς. Οι εταιρικέ σχέσεις δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν πελάτες, έχουν υπηκόους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως αυτός ο επικισμός είναι ε, γεγονός και δεν πρέπει να τον ξεχνάμε, ιδιαίτερα όταν ε, γίνεται λόγος για το κινηματογράφο. Τώρα, ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι κάτι το εκπληκτικό ακριβώς γιατί χαρακτηρίζεται από τεράστια πολυμορφία. Είναι πολύ πλούσιος. Έχει μεγάλη ιστορική παράδοση. Για μένα τα μεταποτε... Ε, ο μεταπολεμικός Ιταλικός κινηματογράφος, η δεκαετία ε, του 60 στην Τσεχία, ο Γαλλικός κινηματογράφος, όλοι ο Ισπανικός έχουν δώσει εκπληκτικές ταινίες, σκανδιναβικό κινηματογράφο, βέλγικος, γερμανικός. Υπάρχουν ταινίες από όλη την Ευρώπη. Όλες είναι διαφορετικές, όλες έχουν διαφορετικό ύφο, ακολουθούν διαφορετική παράδοση, δίνουν έμφαση σε διαφορετικά θέματα. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Αυτό πρέπει να υπερασπιστούμε. Και θα ήθελα να πω κάτι, χωρίς να σταθώ πολύ σε αυτό, ότι σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πω ότι η στήριξη στον κινηματογράφο είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ιδέες, όμως υπάρχει περιορισμός. Υπάρχει αυτό που λέγεται Creative Europe, υπάρχει το Ταμείο για τα Μέσα, το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχουμε ωφεληθεί ως ε, χώρα από αυτό. Το Creative Europe έχει στηρίξει σενάρια, βρετανικά σενάρια και αυτό θα εξαφανιστεί όταν αποχωρήσει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πιστεύω πως θα έπρεπε να συνεχίσει να στηρίζει τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Υπάρχει στήριξη και ε, μέσω χρηματοδότησης. Και εδώ η χώρα μας συμμετείχε. Βέβαια η συντηρητική κυβέρνηση το 1995 μας έβγαλε από αυτό το πρόγραμμα και αυτό, γι' αυτό είναι υπεύθυνοι. Τώρα όμως τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να τους παρακαλέσουμε για να επιστρέψουμε. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να καταστραφεί ο κινηματογράφος της χώρας μου. Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί, πολλοί σκηνοθέτε οι οποίοι θα προσχωρήσουν σε αυτές τις νέες συμφωνίε ή για φορολογικού λόγους. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τις ε, συγκεκριμένες συνθήκες. Υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις για παράδειγμα με το Βέλγιο. Έχουμε εργαζόμενους Βέλγους που δουλεύουν σε βρετανικές ταινίε και είναι πάρα πολύ καλό αυτό γιατί μας φέρνουν βέλγικη σοκολάτα, μας φέρνουν την παράδοση του Ζακ Μπρέλ, τη μουσική, μας φέρνουν πολλά θετικά στοιχεία και είναι πολύ καλή η συνεργασία μας. Όμως η συμπαραγωγή Βρετανίας και Βελγίου λειτουργεί ακριβώς γιατί ευνοεί τη συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής. Όμως, για να έρθουν σε εμά πρέπει να συμπληρώσουν διάφορα γραφειοκρατικά έντυπα και αν δεν το κάνουν δεν θα συμβεί δεν θα γίνει ταινία, θα αποτύχει όλη αυτή η συμπαραγωγή. Αυτά λοιπόν είναι τα άσχημα νέα. Τώρα, υπάρχει τεράστιο πολιτισμικό όφελος ε, όταν συνεργάζεσαι με άτομα από άλλες χώρες, ε, κάνεις φιλίες, βλέπεις τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Σίγουρα αυτό είναι αμοιβαία ωφέλιμο και Σίγουρα το να υποχωρήσουμε στη δική μας εθνική σπηλιά είναι κάτι το πάρα πολύ επιζήμιο. Και σκεφτόμουν πάρα πολύ αυτά που θα πω σήμερα και σκέφτηκα και μία φήμη που κυκλοφορεί ότι κάποιοι Ευρωπαίοι επίτροποι θέλουν η Ευρώπη να είναι μία ενιαία οντότητα ως, ε, σε ό,τι αφορά τις πωλήσει των ε, ταινιών. Και αυτό είναι χαζό. Πείτε μου πως δεν είναι αλήθεια. Και πιστεύω πως είναι χαζό γιατί θα είναι επιζήμιο ακριβώς για αυτή την πολυμορφία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Όταν ε, θεωρείς τα πάντα ως ένα ενίο σύνολο, πώς θα προστατεύσεις τη, την τσέχικη γλώσσα, πώς θα προστατεύσεις τον, βελγικό κινηματογράφο, πώς θα προστατεύσεις τη γλώσσα που είναι συνειφασμένη με την ιστορία μιας χώρας. Δεν μπορούμε να βάλουμε όλα αυτά μαζί στο ίδιο καζάνι και να βγάλουμε μία ευρωπαϊκή άμορφη μάζα. Θα είπα νωρίτερα ότι θέλω να μιλήσω για το Βρετανικό δημοψήφισμα και γι' αυτό το μαρτύριο που έχουμε τραβήξει από τότε. Καταρχάς υπάρχει και ένας μύθος που θέλω να διαψεύσω πολλοί μου λένε ότι η Βρετανία ψήφισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η εργατική τάξη χαρακτηρίζεται από ρατσισμό. Αλλά τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Δύο τρίτα των ψήφων υπέρ της αποχώρησης ήρθαν από το Συντηρητικό Κόμμα, ένα τρίτο από το Εργατικό Κόμμα και κατανοητό αυτό προήλθαν από περιοχές όπου οι παλιές βιομηχανίες έχουν εξαφανιστεί, όπου τίποτα δεν είναι όπως πριν, όπου υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν με συμβάσεις μηδενικών ορών, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, χαρακτηρίζεται από επισφάλεια η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων, οι πολιτικοί δεν τους ακούν, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες και ό,τι και αν ε, λένε, οι πολιτικοί κάνουν το αντίθετο. Από εκεί λοιπόν ήρθαν και όλες οι ψήφοι υπέρ της αποχώρησης, αλλά υπεύθυνη γι' αυτό είναι η δεξιά στη χώρα μου. Η αριστερά όμως είχε και εκείνη ένα δίλημα. Και μιλώ για τη σοβαρή αριστερά και όχι για τη σοσιαλδημοκρατική αριστερά. Η σοβαρή αριστερά λοιπόν είχε ένα δίλημα. η αληθινή ας πούμε αριστερά. Και το δίλημα ήταν το εξής. Θέλουμε να παραμείνουμε σε έναν οργανισμό δεξιό, βασισμένο στην εξουσία των επιχειρήσεων ή αποχωρούμε και όχι μόνο αφήνουμε πίσω μας όλους τους συμμάχους που θα πολεμούσαν στο πλευρό μας, αλλά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια Βρετανική κυβέρνηση η οποία είναι πιο δεξιά από οποιαδήποτε δεξιά κυβέρνηση στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το δίλημα. Ήταν ένα ζήτημα τακτικής, αν θέλετε, γιατί ο εχθρός βέβαια είναι ο νεοφιλελευθερισμός και το θέμα είναι πώς θα τον καταπολεμήσεις και από μέσα και εξωτερικά. Όμως πιστεύω ότι από αυτά που άκουσα, από αυτά που είδα στην Ευρωπαϊκή Τηλεόραση, από τους Ευρωπαίους ε, ηγέτες, είναι ότι δεν εισακουστήκαμε. Αυτό που ακούω είναι ότι το ερώτημα είναι θέλουμε την ανεξαρτησία μας ξανά ή θέλουμε να είμαστε υπήκοοι των γραφειοκρατών στις Βρυξέλλες. Ήταν τόσο βλακώδες το ερώτημα. Τόσο πεδαριώδες. Όμως, το τι Ευρώπη θέλουμε να έχουμε, το οποίο είναι και το σοβαρό ερώτημα, το πώς θέλουμε να είναι αυτή η Ευρώπη, το αν θέλουμε να ζει ο ένας δίπλα στον άλλον με αξιοπρέπεια, το αν θέλουμε μια Ευρώπη όπου όλοι θα έχουν δουλειά, όλοι θα έχουν ένα μισθό για να ζήσουν τις οικογένειές τους, όλοι θα συμπεριφέρονται στον συνάνθρωπό τους ως άνθρωπο. Αυτό, αυτή είναι μια συζήτηση που δεν έγινε ποτέ. Και η αριστερά αντιμετώπισε αυτές τις δυσκολίες γιατί, και θα σας πω ακριβώς όπως τα σημείωσα, ε, δηλαδή, ας κοιτάξουμε τις συνθήκες, τι ιδρυτικές συνθήκες, τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 119. Τα κράτη απαιτείται να εγκρίνουν οικονομική πολιτική η οποία θα διεξάγεται σύμφωνα με την οικονομία της ανοιχτής αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού του. Άρθρο 120 λέει ότι τα κράτη θα πρέπει να ε, ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Αυτά δεν είναι απλές λέξεις. Αυτά τώρα έχουν εξαπλωθεί σε κάθε πτυχή της οικονομίας της Ευρώπης και δεν τα ήξερα μέχρι που το έψαξα ότι υπάρχει και κάτι που ονομάζεται τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Εσείς ενδεχομένως είστε ειδικοί γι' αυτό, εγώ δεν το ήξερα. Αυτό όμως το πακέτο αποτρέπει να περάσει η ιδιοκτησία των συνδυνοδρόμων πίσω στα χέρια μας, πίσω στο δημόσιο. Παραμένει σε ιδιωτικά χέρια. Αν έχει ένα εισιτήριο για μία εταιρεία, δεν μπορεί με αυτό το εισιτήριο να πα σε ένα τρένο άλλη εταιρεία, γιατί υπάρχει αυτή η ιδιωτικοποίηση. Ενώ κάποτε υπήρχε ένα εισιτήριο, οι συντηρόδρομοι ήταν δημόσιοι, με όλα τα προβλήματα που είχαν. Υπήρχαν προβλήματα. Όταν όμως έγινε η ιδιωτικοποίηση υπήρξαν ατυχήματα, υπήρξαν θάνατοι και αυτό γιατί η κάθε εταιρεία έριχνε το φταίξιμο στην άλλη. Έριχνε αλλού τις ευθύνες. Όμως το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο απαιτεί όλα τα κράτη-μέλη να ανοίξουν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην ιδιωτική αγορά. Επίσης αναφέρεται στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, στο ρεύμα, στο νερό. Εσείς τι έχετε στις χώρες σας, Ποιου ποιους παρόχους νερού έχετε στις χώρες σας, είναι ιδιώτες, είναι το δημόσιο. Τι γίνεται με τη στέγαση. Αφήστε με να σας πω κάποια πράγματα με τη στέγαση. Η στέγαση αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε τόσο άσχημη κατάσταση που υπάρχει κόσμος που είναι άστεγος. Η TTIP είναι μια τελειωμένη, αποτυχημένη συμφωνία. Όχι, αν δεν κάνω λάθος υπάρχει μια αντίστοιχη συμφωνία με τον Καναδά όπου οι επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις λοιπόν θα είναι υποχείρια των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Είμαστε σοβαροί. Αυτά σκέφτονται στην Ευρώπη. Και φυσικά η αριστερά, δεδομένων όλων αυτών, σκέφτεται πως καλύτερο είναι να αποχωρήσει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης υπάρχουν και πολλές αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες περιορίζουν τη δύναμη των συνδικάτων, περιορίζουν την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων. Δεν είναι λάθος όλα αυτά. Υπονομεύουν τους εργαζόμενους. Πώς μπορείτε λοιπόν να στηρίζετε κάτι τέτοιο, πώς μπορείτε να στηρίζετε την υπονόμευση της εργατικής τάξης. Αυτό είναι λοιπόν το δίλημα. Το γεγονός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στην ιδεολογία της, έχει στην ιδρυτική της πράξη αυτή την νεοφιλελεύθερη ατζέντα. Είναι γραμμένο παντού. Είναι ένα σύνθημα, είναι ένα αυτοκόλλητο σε κάθε σελίδα. Βρίσκεται στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ πως είναι μία πάρα πολύ άσχημη ένωση για την εργατική τάξη. Ήταν λοιπόν μια απόφαση πιο πολύ στρατηγικής. Θεωρώ πως Είμαστε, ε, θεωρώ πως είστε ε, περήφανοι λοιπόν για τα αποτελέσματα αυτά, για ανεργία πάνω από το 10%, για ανεργία των νέων που σε ορισμένες περιπτώσεις πλησιάζει το 50%, την άναδο της ακροδεξιάς, την άναδο του ρατσισμού. Ο Νάιτζελ Φαράς ε, αυτή τη στιγμή έχει δουλειές για τι έχει δουλειά στο να απασχολούν οι αμερικανικέ εκλογέ και το τι γίνεται με τον Ντόναλτ Τραμπ. Λείπει λοιπόν, αλλά εάν ψάξουμε για ε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ας δούμε τι έχει γίνει στην Ελλάδα, ας δούμε τι έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. Είναι έχουν ένα χρέος το οποίο δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποπληρώσουν και αναγκάζονται να ξεπουλήσουν την δημόσια περιουσία. Γιατί προ όφελο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες θέλουν να καταλυστέψουν τον ελληνικό λαό, να πάρουν ό,τι υπάρχει. Δεν υπάρχει λοιπόν καθόλου καλό ιστορικό. Και τώρα περνάμε στα νέα από τη Βρετανία. Στη Βρετανία Έχουμε μια κοινωνία που είναι ε, σκληρή, αποξενωμένη, εξαγριωμένη και διαιρεμένη. Ναι, έχουμε ακόμη μαζική ανεργία, αλλά έχουμε 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι στη μερική απασχόληση. Ενδεχομένως δουλεύουν μία-δύο μέρες την εβδομάδα που δεν είναι τμήμα των στατιστικών της ανεργίας, αλλά πραγματικά χρειάζονται χρήματα από το κράτος για να επιβιώσουν. 5,5 εκατομμύρια μερικώς απασχολούμενοι με συμβάσεις ε, μηδενικών ορών, ε, ε, με, απασχόληση, με απασχόληση κατά την οποία μπορεί να δουλεύεις μία μέρα, δύο μέρες, αλλά όχι την υπόλοιπη εβδομάδα. παρόλα αυτά πρέπει να είσαι διαρκώς διαθέσιμος. Μίλησα για τους άστεγους, μίλησα για το πρόβλημα της στέγασης. Στο Λονδίνο, όπως γνωρίζετε, ε, άνθρωποι, εργαζόμενοι δεν μπορούν να βρουν πού να μείνουν στο Λονδίο γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά τα ενίκια. Μιλούσα σε έναν δάσκαλο δημοτικού πριν από δύο μέρες που έπρεπε να φύγει το, από το Λονδίνο και είναι ε, μίλια μακριά γιατί δεν μπορεί να ζει στο Λονδίνο. παράλληλα, ε, τα κτηματομεσητικά, η αγορά κινήτων, ε, οικοδομή ε, τεράστια, ε, τεράστιες ε, πολυτελείς πολυκατοικίες που το βράδυ δεν έχουν φώτα γιατί, γιατί κανείς δεν μένει μέσα και γιατί, γιατί ήταν απλώς επενδύσεις 50 εκατομμύρια λίρες ε, κάνουν ε, τα διαμερίσματα στο Λονδίνο. Αυτή είναι η αγορά. Αυτή είναι η αγορά κινήτων ε, στο Λονδίνο. Οι πυροσβέστες, οι νοσοκόμες, οι δάσκαλοι δεν μπορούν να ζήσουν μερικά χιλιόμετρα στην περιοχή, γύρω από την περιοχή όπου εργάζονται. Και να ολοκληρώσω σιγά σιγά. Μία ερώτηση και πιστεύω ότι κάποιος θα ξέρει την απάντηση από εσά, σίγουρα. Έχουμε, είμαστε μια χώρα τεράστιων ε, ανισοτήτων, ε, ε, έχει πέσει κατά 50% ε, ε, έχει ανέβει κατά 50% συγγνώμη, ο μισθός των νότατων στελεχών κατά την κυβέρνηση των συντηρητικών και έχει μειωθεί του μέσου εργαζόμενου. Σε 45 λεπτά μπορεί ένα νότατο στέλεχος μιας επιχείρησης να κερδίσει αυτά που χρειάζεται ένας μέσος εργαζόμενος ολόκληρο το χρόνο. Αυτό το έκαναν οι συντηρητικοί. Μιλάμε για τεράστιες ανισότητες. Ε, επίσης ε, έχουμε ανθρώπους που δεν τρώνε εκτός εάν κάποιος ε, σε ένα σούπερ μάρκετ ε, βάλει μέσα σε ένα κουβαδάκι που έχουν μπροστά τους κάτι για να φάνε. Είναι ένα πρόβλημα που δεν το είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Και 1,1 εκατομμύρια γεύματα, πακέτα γευμάτων δόθηκαν ε, πέρσι ε, πάνω από 500.000 σε παιδιά. Επίσης η ε, κοινωνική φροντίδα, η φροντίδα των ανθρώπων με αναπηρίες, οι οποίοι, δουλεύουν, οι οποίοι υποφέρουν έξι φορές περισσότερο λόγω των περικοπών. Όταν ακούς ε, λοιπόν την Τερέζα Μέη να ε, λέει ότι είναι, ε, το κόμμα της είναι το κόμμα ε, το, της εργαζόμενης τάξης, πρέπει να σκάτε στα γέλια. Οι πλέον ευάλωτοι έχουν γίνει ακόμη πιο ευάλωτοι. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται πάρα πολύ υποστήριξη, άνθρωποι που είναι πολύ άρρωστοι για να δουλεύουν, όμως τους λένε ότι πρέπει να δουλεύουν. Αυτό πραγματικά είναι μια συνειδητά πολύ σκληρή απόφαση ε, σου λένε ότι αν είσαι φτωχό, εσύ φταίει. Αν δεν έχει ένα σπίτι, εσύ φταίει. για παράδειγμα, υπήρχε μία ε, ιστορία ενός ε, ανθρώπου που έπαθε καρδιακή προσβολή και δεν μπορούσε να δουλέψει. Κατά την αξιολόγησή του για να αποφασιστεί αν μπορούσε ή όχι να δουλέψει έγινε είχε καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αυτής για την αξιολόγηση. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη συνέντευξη, οπότε ε, του επέβαλαν ε, κυρώσεις γιατί δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αξιολόγηση παρά το γεγονός ότι έπαθε καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αυτής. Αυτή είναι η πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες, για εκατομμύρια ανθρώπων. Είμαστε λοιπόν περήφανοι από την, ε, για την κατάσταση αυτή, για την εξέλιξή μας, η νεοφιλελεύθερη Βρετανία και η νεοφιλελεύθερη Ευρώπη. Όχι. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο ε, των έργων μας και η δική μας ευθύνη είναι να λέμε την αλήθεια. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Ε, και κάτι ακόμη το οποίο θα ήθελα και το οποίο μπορεί να προκύψει από τις ερωτήσεις ε, είναι ότι ο νέος ε, ηγέτης των εργατινών ε, για πρώτη φορά, στη για πρώτη φορά στην ιστορία του εργατικού κόμματος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων γιατί θα περιορίσει το θα, θα, θα, περιορίσει ε, τις ε, ε, τις, ε, τις ε, απεργίες. Σκεφτείτε το, οι εργατικοί η εργατικοί στο παρελθόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν υποστηρίξει τους εργάτες όταν, ήταν, όταν μιλούσαν για τις απεργίες. Η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό θα δείτε, θα είναι και η μοναδική φορά που κανείς δεν θα πει κουβέντα για αυτόν στο Βρετανικό τύπο και Δείτε τι θα γίνει, σας το λέω. Τι θα γίνει όταν ε, αυτός ο άνθρωπος θα το κάνει. Δεν πρόκειται κανείς να μιλήσει για αυτόν, γιατί είναι μια πραγματική πρόκληση. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας έχω στο μυαλό μου διάφορες ε, παραθέσεις ε, ανθρώπων που θεωρώ μερικές φορές ότι είναι ένα καλό μότο για όσους ε, κάνουν κινηματογράφο, για τους σεναριογράφους, για όσους προσπαθούν να συμμετέχουν σε αυτήν την τέχνη. Είναι από τον Μπρέχτ, είναι πολύ κακή η μετάφραση και συγγνώμη από τους Γερμανούς για την κακή αυτή μετάφραση. Είχε πει Πάντοτε πίστευα ότι οι απλούστερες λέξεις πρέπει να αρκεί. Όταν λέω ε, πώς είναι τα πράγματα, θα ε, στεναχωρηθούν όλοι ε, το ότι θα χαθεί κανείς αν δεν αγωνιστεί. Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές σε εσά. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε για αυτή την ομιλία σας γεμάτη έμπνευση. Σας δώσαμε λοιπόν τον κατάλληλο χώρο για να ε, πείτε αυτά που είπατε και είπα και πριν, ότι καθήκον των σκηνοθετών, των δημιουργών είναι να λένε την, την αλήθεια. Και εσείς με μεγάλη ελευθερία και μεγάλο στένος μας εκφράσατε τους λόγους ε, οι οποίοι θα πρέπει να μας ε, κάνουν να υποστηρίζουμε αυτή την ελευθερία της έκφρασης των δημιουργών και να σταθώ σε αυτό το πρώτο που είπατε. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας πιο συγκεκριμένα δίνουμε μάχη ώστε να μην προστατεύουμε απλώς ε, την ε, ελευθερία των δημιουργών και να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση ε, στα θέματα αυτά από πλευρά των ανθρώπων, αλλά και για να αναγνωρίζεται και η πολιτιστική ποικιλομορφία ως πλούτος, αλλά και ε, φυσικά να δημιουργήσουμε ένα χώρο πολιτισμού, κινηματογραφίας, ε, της πολιτιστικής βιομηχανίας Ευρώπης που να έχει να πει κάτι στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν θέλουμε ε, να ομογενοποιήσουμε τα πράγματα και να μας επιβάλλουν οι νόμοι της αγοράς τι θα γίνει. Και αυτή η ισορροπία στην οποία αναφερθήκατε είναι το μεγάλο στίχημα του σινεμά και του σινεμά. Είπατε κάποια πράγματα σκληρά, πολύ ισχυρά, με κάποια προσωπικά συμφωνώ, με κάποια άλλα όχι. Εγώ ε, πιστεύω ότι η φιλοσοφία της συνθήκης της Ευρώπης είναι μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, όχι οικονομικός νεοφιλελευθερισμός. Και νομίζω ότι αυτό το καταδεικνύουν πολλές ερμηνείες που δίνουν κάποιες από τις πολιτικές μας ομάδες και για τις οποίες δίνουν και τις μάχες τους. Εσείς αναφερθήκατε στο θέμα της απόσπασης των εργαζομένων και ε, ε. νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει σαφέστατα την άποψή του και ζήτησε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, φροντίσει να υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολείται με την καταπολέμηση της ένδυας. Επομένως, ο καθένας με τις ευαισθησίες του, η πολιτικέ ομάδες έχουν διαφορετικές πολιτικές ευαισθησίες, αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συζήτηση αυτή είναι ανοιχτή. Υπάρχει Φυσικά η άποψη του καθενό, αλλά το συμμεριζόμαστε, γνωρίζουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένη πρόκληση και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αλληλέγγυοι, να προσπαθήσουμε να ε, έχουμε μια ε, σύμπνοια μέσω μιας νέας ευημερία και μέσω μιας νέας ανάπτυξης και να δώσουμε νέα προοπτική και ελπίδα στις νέες γενιές. Οι αδικίες βέβαια που καταγγέλλεται είναι αδικίες τις οποίες γνωρίζουμε, που υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι η ε, κατάλληλη πολιτική, η υψηλή πολιτική θα πρέπει και να τις αναγνωρίζει αλλά να έχει και τη δυνατότητα να τις ξεπεράσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εχθρική στάση στην Ευρώπη. Ε, υπήρχε μια στιγμή στην οποία είχαμε μια ε, νέα ε, ενιαία φιλελεύθερη πολιτική αλλά αυτή τη στιγμή τα ξεπεράσουμε. Νομίζω ότι όλοι μάθαμε το μάθημά μας και ακόμα και αυτοί που δεν συμφωνούσαν ούτω ή άλλω. Δεν θέλω να συνεχίσω εδώ, δεν θα ήθελα να κάνω συζήτηση για τι πολιτικέ σα τοποθετήσει. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που είπατε. Χρειαζόμαστε έναν μάρτυρα ο οποίο θα είναι απαιτητικό, ανυπόμονο και ίσω και άβολε κάποιε φορέ που μα λέει πράγματα που ίσω δεν θέλουμε να ακούσουμε. Σα ευχαριστώ λοιπόν για τα όσα μα είπατε και να δώσουμε το λόγο στην Τόρι Πακ, να την ευχαριστήσουμε που είναι εδώ. Με την Τόρι ε, έχουμε πολλά κοινά ε, σημεία στη ζωή του βραβείου Λίουξ ε, και στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Θα της δώσω το λόγο λοιπόν για να πει δυο λόγια και να δώσει στη συνέχεια το λόγο ε, στους άλλους δύο σκηνοθέτε μας, τους οποίους έχουμε προσκαλέσει εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνώρισα τον Κέν Λότς πριν από πέντε χρόνια και δεν άλλαξε καθόλου πριν από πέντε χρόνια μου εξήγησε τον σοσιαλισμό σε ένα δείπνο μαζί με τη γυναίκα του. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά και συμφωνήσαμε σε όλα όσον αφορά τον σοσιαλισμό και τους σοσιαλιστές. Ε, γι' αυτό λοιπόν δεν νομίζω πως εδώ χρειάζεται να διαφωνήσουμε. Ε, όμως πιστεύω πως δεν πρέπει να ρίχνουμε το φταίξιμο στην Ευρώπη για όλα. Θα ήθελαμε λοιπόν μαζί με τον Κέν Loach να ε, δώσουμε την αφορμή να ανοίξει μια συζήτηση για το τι πρέπει να βελτιωθεί. Πολλές φορές βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως ε, τα θέλουμε από την προσωπική μας σκοπιά. Όμως εκτός από τον πολύ σημαντικό Ken Loach έχουμε και δύο άλλους σημαντικούς ανθρώπους, την ε, Σελήνη Σαμά που έκανε αυτήν την εξαιρετική ταινία «Τα κορίτσια» και τον Αντρέ Σέγκρε, ο οποίος έχει κερδίσει το βραβείο Λουξ με την ταινία «Εγώ ήσουν Είδα ε, το, την ταινία του Ken Loach, το εγώ Daniel Blake στις Κάνες ε, και πρέπει να πω ότι αυτές είναι ταινίες που ασχολούνται με πολύ σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Δυστυχώς όμως ε, οι ταινίες είτε είναι ιταλικές, γερμανικές, εστονικές είτε οτιδήποτε άλλο όταν είναι σε μια γλώσσα εκτός από ε, αγγλικά είναι δύσκολο να τις καταλάβουμε. Γι' αυτό λοιπόν και δημιουργήθηκε το βραβείο Lux. Οι ταινίε παρουσιάζονται, υπάρχει μια κριτική επιτροπή η οποία επιλέγει τρεις και η κριτική επιτροπή δεν αποτελείται από ευρωβουλευτές, αποτελείται από ειδικού και μετά επιλέγονται λοιπόν οι τρεις φιναλίστ και εμείς τις ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για τον νικητή. Το θέμα όμως είναι να μπορέσουμε να δούμε αυτές τις ταινίες. Η ταινία του Ken Loach δεν φαντάζομαι να έχει ένα τεράστιο κοινό. Ακριβώς γιατί η ταινία του στέλνει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα και είναι μια πολύ συγκεκριμένη ταινία. Και εάν δεν υποτιτλιστεί είτε στα γερμανικά, είτε στα γαλλικά, είτε στα πολωνικά, δεν θα τη δει πολλοί κόσμος, θα τη δει ακόμα λιγότερος ε, κόσμος. Τώρα, κυρία Σέρμα να πω ότι δημιουργήθηκε και στου κινηματογράφου. Είτε επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα διανομή, είτε επειδή δεν έχουν υποτιτλιστεί. Είναι όμω μια πλατφόρμα που δημιούργησε η κυρία ε, Σαμά για αυτέ τι ταινίε. Θα μπορούσατε να μα πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, δεν είναι μόνο εκπαιδευτική ε, πλατφόρμα. Είναι μια πλατφόρμα VOD, είναι κάποιο είδους σινεματέκ, ε, βιβλιοθήκη κινηματογράφου ε, με σκηνοθέτες, σεναριογράφους, είναι, έχουμε τέρους πάρα πολλούς και ε, στη Γαλλία και η ιδέα ήταν ε, να, υπάρχουν, να υπάρχει συγκέντρωση ε, ε, ταινιών του 20ου αιώνα ε, παράδοσης ε, επιλέγονται και γίνεται μία διαμόρφωσή τους από κάποιους σκηνοθέτες. Ίσως και ο Κεν Λαούτς να μπορούσε να μας δώσει έναν κατάλογο. 50, 50 ταινίες προτείνει κάθε σκηνοθέτης οι οποίες θα αναδιαμορφωθούν και θα συγκεντρωθούν. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να βρεθούν αυτές ε, οι ταινίε. Ε, ούτε είναι και πάρα πολύ δύσκολο πάντα, αλλά είναι διασκορπισμένες από εδώ και από εκεί και η ιδέα είναι να να αποφασίζουν ε, οι σκηνοθέτες που θα μιλούν για τις ταινίες τους αυτές. Υπάρχει λοιπόν μία τέλο πάντων εκπαιδευτική αξία παρουσίασης αυτών των ταινιών και κάποιων σχολείων που θα τη συνοδεύουν. Όμως, Ελπίζουμε να επεκταθεί και στην Ιταλία και στο Βέλγιο. Για κάθε φορά πρέπει να γίνεται η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων. Δεν είναι εύκολο. Αν πάση περιπτώσει είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, δεν είναι ακριβώς ε, αγορά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, για την ώρα δεν υπάρχει οικονομικό μοντέλο. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να την υποστηρίξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σελήν. Θα ήθελα και να ρωτήσω τον Αντρέ κάτι παρόμοιο. Από όσο ξέρω, έχετε μεγάλο ενδιαφέρον για τα ντοκιμαντέρ. Ε, και δυστυχώς, ε, οφείλω να ομολογήσω ότι τα ντοκιμαντέρ δεν ε, έχουν τόσο μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό όσο οι άλλες ταινίες οι ταινίε μυθοπλασία. Και έχετε δημιουργήσει κι εσεί μια ανεξάρτητη εταιρεία η οποία επιτρέπει στου θεατέ να βλέπουν ε, δωρεάν ντοκιμαντέρ. Μπορείτε να μα πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Ναι. Ευχαριστώ. Πράγματι, αυτό δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση από καλλιτεχνικής απο, απόψεως. Πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με ένα κοινό που είναι ε, βασικά νέοι. Νομίζω ότι η απόσταση μεταξύ της φαντασίας και του ντοκιμαντέρ είναι πάρα πολύ ωραία και πρέπει να γίνεται αυτή η απόσταση. Υπάρχουν ε, πραγματικοί άνθρωποι που γίνονται εξαιρετικοί ηθοποιοί και πραγματικοί εξαιρετικοί ηθοποιοί που γίνονται πραγματικοί άνθρωποι. Και οι ιστορίε που παίρνουμε εμεί από την πραγματικότητα είναι αυτέ οι οποίε μα επιτρέπουν στη συνέχεια να δημιουργηθούμε ιστορίε οι οποίε ε, ε, στέκονται μπροστά στην πραγματικότητα αλλά μπορούν να πάνε και πέρα από αυτήν. Το πρόβλημα βέβαια είναι να προβληθούν αυτέ οι ιστορίε. Και Πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα έχει και μεγάλη σχέση με αυτά τα οποία μας διηγήθηκε ο Κεν Λόουτς, όχι μόνο για τον κόσμο του σινεμά, αλλά και για το οικονομικό σύστημα το οποίο, στο οποίο ζούμε. Υπάρχει μια τεράστια ανισότητα και στην αγορά της ε, διανομής ε, κινηματογραφικών ταινιών, ε, η οποία σχετίζεται και με τη δυτή ταυτότητα του κόσμου του σινεμά. και της βιομηχανίας, ε, τα οικονομικά συμφέροντα ορισμένες φορές ε, έχουν σχέση όχι μόνο με την παραγωγή αλλά και τη διανομή των ταινιών. Εγώ δεν είμαι πολύ καλός ε, στις ομιλίες. Αυτό που κάνω στη ζωή είναι να διηγούμε ιστορίες και θα σας διηγηθώ μια ιστορία για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Θα σας πω μια ιστορία στην οποία δεν μπορώ να σας πω τα ονόματα των πρωταγωνιστών διότι ε, όχι μόνο γιατί δεν του ζήτησα την άδεια αν μπορώ να διηγηθώ την ιστορία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχω το ελεύθερο, αλλά ε, γιατί για αυτούς θα ήταν πολύ δύσκολο να την πουν δημοσίως αυτή την ιστορία. Είναι η ιστορία δύο νέων παιδιών που τους τελευταίους μήνες ε, έσωσαν μια κινηματογραφική αίθουσα σε μια μικρή κομμόπολη 10.000 κατοίκων στην Ιταλία. Ήδη πρέπει να τους στήσουμε άγαλμα, γιατί το να διασώσουν στα 28 του μία αίθουσα κινηματογράφου είναι ένα τεράστιο πολιτιστικό εγχείρημα. Και το έκαναν από πάθος, γιατί τους αρέσει το σινεμά. Δεν υπάρχει άλλος λόγος, κάνουν διαφορετική δουλειά. Ο ένας είναι λογιστής και ο άλλος είναι γραμματέας ε, σε κάποιο ε, γραφείο λογιστών. Αλλά ε, τους αρέσει το σινεμά και διέσωσαν μία αίθουσα κινηματογράφου που έκλεινε και η περιοχή, η ενορία, γιατί ήταν η αίθουσα του κινηματογράφου τη να την κλείσει γιατί δεν έβγαζε πια χρήματα. Και είπαν όχι θα τη σώσουμε και άρχισαν να εργάζονται δωρεάν για να σώσουν την κινηματογραφική αίθουσα. Την έσωσαν και μετά είπαν ωραία τώρα που τη σώσαμε μετά από τις προσπάθειές μας να κάνουμε ε, μια εκστρατεία στην πόλη, να προσπαθήσουμε να συμμετέχουν κι άλλοι και ε, να, με μια ευκαιρία πώς τη λέμε σήμερα, sharing economy, να μοιραζόμαστε και να υπάρχει συμμετοχή από όλε τι πλευρέ. Ε, είπανε ωραία, έχουμε την αίθουσα, την ε, έφτιαξαν και λίγο, βάλανε και νέο προβολέα, ε, έχουμε την αίθουσα, μπορούμε να μείνουμε ε, όσο μα αρέσει γιατί μα αρέσουν και οι ταινίε. Και άρχισαν να σκέφτονται να υπάρχει και πρόγραμμα ταινιών για το, την κινηματογραφική αίθουσα. Είναι και γονεί, έχουν παιδιά και τα παιδιά του τους είπαν, ναι, αλλά μπομπά να ε, δείξουμε και την ταινία του Walt Disney που μόλις βγήκε. Ναι, βεβαίως. Κάλεσαν τον Ιταλό διανομέα της ταινία, ε, το ταξίδι της Ντόρι, μία που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ε, αυτά τα ονόματα μπορώ να σας τα πω, τα άλλα όχι. Τηλεφώνησαν λοιπόν στο διανομέα και ο διανομέας τους είπε βεβαίω. θέλετε την ταινία μας. Πολύ ωραία, ναι, ναι, θέλουμε, θέλουμε να την προβάλλουμε Σάββατο και Κυριακή το απόγευμα ε, ως οικογενειακή ταινία. Αν θέλετε να το προβάλλετε Σάββατο και Κυριακή πρέπει να το δείξετε και Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ, κάθε Τρίτη, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη για κάθε βράδυ για τρεις εβδομάδες. Αλλιώς 5.000 ευρώ πρόστιμο. Ε, μα εμείς θέλουμε να προβάλλουμε Σάββατο και Κυριακή την ταινία και μετά στη διάρκεια της ημέρας δείχνουμε ντοκιμαντέρ, έχουμε καλέσει και τον Αντέα Σέγκρε με τον ντοκιμαντέρ του, δεν καταλάβαμε τι μας είπατε. Εάν θέλετε να δείτε την ταινία πρέπει να σεβαστείτε αυτή τη συμφωνία. Τελικά καταφέρανε να δείξουν το ντοκιμαντέρ μου μια Τετάρτη βράδυ και πήγα και του συνάντησα κιόλα και μου διηγήθηκαν αυτή την ιστορία και του είπαν ναι, βεβαίω, δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούω αυτό. Και με ρώτησαν κάτι πολύ απλό, το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ σε εσά γιατί δεν υπάρχει ένας χώρος στον οποίο εμείς να μπορούμε να καταγγείλουμε αυτό το γεγονός, διότι πρόκειται περί Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι λάθος να με υποχρεώνεται να ε, δείχνω μια ταινία βάσει μιας οικονομικής συμφωνίας η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο θέλει να δει ο κόσμος στο σνεμά μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χώρο στον οποίο ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα, διότι έχουν σχέση με άλλες ανισότητες, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τον κόσμο του σινεμά ε, αυτά τα χρόνια με τις ταινίε μου διέσχισα την Ιταλία προσπαθώντας να βοηθήσω αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν αίθουσες κινηματογράφου και ο καθένας δίνει μια άνηση μέχη. Ε, ορισμένες φορές υποχωρούν, διότι αν κάποια στιγμή δεν σε βοηθάει κανείς αυτή τη μάχη κατά το γραφείο της Fox ή της Walt Disney, ε, που προφανώς είναι ένας τηλεφωνικός αριθμό στον οποίο καλείς και σου επιβάλλει απλώ κανόνε, ταινία και παύλα. Πώς μπορείς να βοηθήσεις το κινημά, το, σινεμά, το διαφορετικό σινεμά να επιβιώσει. Εμείς ε, ε, μπορούμε να έχουμε αίθουσες διανομής, έχουμε ιδέες, αλλά εάν δεν αλλάξουν αυτές οι κανόνες, κερδίζει απλώς η λογική της αγοράς και κανείς άλλος. Αυτή ήταν μια υπέροχη ιστορία και θα ήθελα να συμπληρώσω και να κλείσω λέγοντας ότι όπως είπε και ο Κέν Λόουτς κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν ακριβώς αυτά τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία για παράδειγμα στην Πολωνία χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα για να σώσουν κινηματογράφους, για να ψηφιοποιήσουν κινηματογράφους οι οποίοι βρίσκονταν μακριά από τις πόλεις, δεν είχαν εξοπλιστεί με τη νεότερη τεχνολογία και δεν μπορούσαν να δείξουν, να προβάλλουν τις καινούργιες ταινίε. Να λοιπόν ένας, ε, ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς μπορεί να ενωθεί η ε, οικονομία με την τέχνη. Δεν ε, πρόκειται μόνο και στεγνά για χρήμα, αλλά μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Αυτό θα ήθελα να το πω προς απάντηση στον κύριο Λότς. Επιτρέψτε μου όμως να προσθέσω και κάτι άλλο. Όλες οι ταινίες του Ken Loach, εκτός από την τελευταία, διατίθενται δωρεάν. Όποιος δηλαδή θέλει να τις δει, μπορεί να τις δει δωρεάν. Όλες λοιπόν οι ταινίες του Ken Loach, εκτός από την τελευταία. Και το θεωρώ καλό, αλλά νομίζω πως ε, ο κύριος Loach έχει την πολυτέλεια να το κάνει αλλά ο κύριο Σέγκρε, η κυρία Σαρμά δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια να το κάνουν. Εντάξει, μπορεί να είναι και θέμα ηλικία, αλλά δεν έχουν όλη αυτή την ε, δυνατότητα. Θα ήθελα όμω να το αναφέρω. Ε, κυρία Πρόεδρε, εσεί όμω ε, θέλετε το λόγο. Λοιπόν, καταρχά, ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Θα ήθελα να πω το εξή στον Αντρέα Σέγκρε, διότι αναφερόνται σε μια ιταλική κατάσταση την οποία γνωρίζω πολύ καλά. Στην Ιταλία μόλι εγκρίθηκε μια νομοθεσία η οποία αναφέρεται στην προστασία των αιθουσών κινηματογράφου ιστορική σημασία ή που έχουν κάποια άλλη μορφή σημασία. Είναι βέβαια γενικευμένο το ζήτημα. Σίγουρα μπορούμε να παρέμβουμε μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείου, αλλά πρέπει να βρούμε και κάποια οικονομικά μοντέλα τα οποία να υποστηρίζουν στη συνέχεια τη διανομή ταινιών ποιότητα Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε κι άλλο και σε κάποιες περιπτώσεις, ε, το ξέρω γιατί το έχω ε, επαληθεύσει, ε, μπορούμε να προτείνουν και κάποιες μορφές μονοπωλίου ή επιβάλλουν κυρώσεις και το καθεξής. Αλλά υπάρχουν και διεθνείς συνομιλητές και υπάρχει και ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να ξέρω αν θέλουν οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο. Ο Κούρτσο Μαλτέζε, η κυρία Τρίπελ καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κεν Λόουτς πάρα πολύ, γιατί μου άρεσε τόσο πολύ αυτός ο φρέσκος και εμπνευστικό σας λόγος, ειδικότερα για το φως, που μερικές φορές μπορεί να είναι ψυχρό ή πολύ ψυχρό και την ανάγκη για ζέστη, για θέρμη. Φαντάζεστε ότι πολλές φορές ε, οι λόγοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι τόσο φρέσκοι, οπότε το, τον απόλαυσα πραγματικά, ε, ειδικότερα όσον αφορά τον κινηματογράφο, το ότι είναι ειδική μορφή τέχνης και το χρειαζόμαστε τόσο πολύ για να στραφούμε προς τους, να πλησιάσουμε τους ε, θεατές και να τους ε, εμπνεύσουμε. Όσον αφορά το γεωγραφικό αποκλεισμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές ταινίε. Απ' την άλλη πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην έχουμε μία ε, άδεια ε, που θα μπορεί να ε, είναι προσιτή μόνο στους Αμερικάνους για παράδειγμα και όχι στους Ευρωπαίους γιατί θα είναι πάρα πολύ ακριβή. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πρόσβασης για τους πολίτες στο ευρωπαϊκό περιεχόμενο όμως δίνοντας τη δυνατότητα διατήρησης πολιτιστικής ποικιλομορφία και δημιουργίας ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Όσον αφορά αυτό που είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα με την κατάσταση στο Βασίλειο, αλλά το να δίνεται την εντύπωση μιας μόνο νεοφιλελεύθερης ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Μπορείτε να επικρίνετε πολλές πολιτικές, όμως υπάρχουν και ρυθμισμένε αγορές. Δείτε την Τραπεζική ε, Ένωση, δείτε για παράδειγμα την πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Γενικώ οι περιβαλλοντικέ πολιτικέ που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των αγορών. Το να δίνεται λοιπόν η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο νεοφιλελεύθερη καταστρέφει σε κάποιο βαθμό ε, την ε, ε, εμπιστοσύνη των ανθρώπων όταν κινούνται συλλογικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχουν, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν πηγαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση, συμφωνώ, αλλά ε, υπάρχει και κάποια θέληση και κάποια ε, επιτυχία από τη ρύθμιση των αγορών και αυτό δεν είναι ε, κακό. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω ότι για λόγους επικοινωνίας πρέπει να βγούμε όλοι Θα αφήσω την Προεδρία στη συνάδελφο στην κυρία Τρούπελ, αν θέλετε να έρθετε στο Προεδρείο, γιατί πρέπει να βγούμε. Ε, είστε αντιπρόεδρος άλλωστε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική αυτή χειρονομία. Σας αφήνω και θα τα πούμε αργότερα στις 7 στο Παρλαμεντάριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Βέντα από την Πολωνία. Ευχαριστώ. Ντόρις, ε, ευχαριστώ που αναφέρθηκες στον ε, κινηματογράφο μας ε, στην Πολωνία που επιβίωσε. Να ξεκινήσω με αυτό που συνέβη εχθές το βράδυ. Ο Άντρεϊ Εβάιντερ δυστυχώς απεβίωσε. Ε, αν λάβει κανείς υπόψη τα 40 τελευταία του έργα, τα οποία είναι γνωστά και διεθνώς, αλλά είναι και πολύ σημαντικά για την Πολωνία, αυτό δείχνει, αυτό από μόνο του δείχνει, πόσο πώς μπορεί κανείς να προωθήσει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο ε, απεικόνιζε όχι μόνο το παρελθόν της δικής μου χώρας Πολωνίας, αλλά ήταν και ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό στοιχείο για την αλλαγή στην Πολωνία. Δεν ήταν μόνο φανταστικός δημιουργός, αλλά ήταν επίσης ένας πολύ καλός δάσκαλος, ε, παιδαγωγός της κοινωνίας μας. Και κάτι ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι όχι μόνο μέσω των διαδοτικών ταμείων, αλλά και μέσω του Creative Europe, οπτικοστικός τομέας, ε, την κάνει υποστήριξη. Εγώ ήμουν εισηγητής ε, όσον αφορά τον κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή και εδώ νομίζω ότι είναι σαφές ότι πρέπει να υποστηρίξουμε το βραβείο Λουξ γιατί προωθεί τις ευρωπαϊκές ιδέες και τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, ειδικότερα σε μια περίοδο κρίσης αξιών και ευρωσκεπτικισμού, όπως, και σε χώρες όπως και η Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ward. Ε, σας παρακαλώ μην αναφερθείτε στο Brexit όμως. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη, σύντομη. Ο Κέν και εγώ ήμασταν στην ίδια πλατφόρμα πριν από μερικές εβδομάδες και μιλούσαμε κατά ε, του κλεισίματος ε, το νοσοκομείο γυναικών του Λίβερπουλ. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Μ' αρέσει πολύ η δουλειά σου. Εγώ δούλευα στον τομέα των τεχνών πριν έρθω εδώ. Ε, και τώρα κατά πόσο είμαστε σοβαροί και πραγματικοί σοσιαλιστές εγώ άφησα πίσω μου μία ζωή στις τέχνες για να πολεμήσω για πράγματα που με ενδιαφέρουν πολύ. Πιστεύω ότι είναι ένας ε, σοβαρός, είμαι μια σοβαρή σοσιαλίστρια ε, και υποστηρίζω τον Τζέρεμι. Χαίρομαι πάρα πολύ για το μήνυμα που είπες, ε, που μας έφερες εδώ. Πολλά πράγματα από αυτά που είπες τα γνωρίζουμε. Τα γνωρίζουμε γιατί τα κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και η δουλειά ενός πολίτη πολιτικού ενός Ευρωβουλευτή είναι στην Επιτροπή. Η δουλειά που κάνουμε εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά ε, πραγματικά πρέπει να βρούμε ε, κοινό έδαφος και συμφωνία με τους εταίρους μας ε, και είναι θλιβερό αυτό που έκανε η χώρα μας ε, είναι να γυρίσει την πλάτη σε αυτή τη συζήτηση γιατί οι πραγματικές αλλαγές μπορούμε να κάνουμε όταν μπορούμε να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι μαζί να συζητήσουμε τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας τη θέρμανση του πλανήτη ζητήματα που συζητούμε και εμείς εδώ και παρά το προβλήματα που έχουμε με με τους ε, εξτρεμιστές. Ε, το κοινοβούλιο έχει περισσότερες γυναίκες, ε, έχει, συγκεντρώνει ανθρώπους που διαφωνούν με ε, με, την φορολογική, ε, με τη φοροαποφυγή. Ε, γίνονται πολλά πράγματα εδώ, περισσότερα από ό,τι στο Westminster και πολλά προβλήματα που βλέπουμε να υπάρχουν στην Ευρώπη, ας πούμε η Ουγγαρία να κλείνει τα σύνορά τη ή ο κόσμος που δεν διασώζει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Είναι μερικές φορές μεμονωμένα κράτη-μέλη, οπότε πρέπει να αγωνιστούμε για την Ευρώπη στην οποία πιστεύουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε πάρα πολλή δουλειά ε, για να ε, μπορούμε να έχουμε εδώ μια πραγματικά αριστερή φωνή. Εγώ θεωρώ ότι είμαι τμήμα αυτή της φωνή, είμαι μέλος των εργανητικών, είμαι μέλος των σοσιαλδημοκρατικών. Όλοι εδώ αγοριζόμαστε, πολεμούμε, ε, πιστεύοντας σε μια Ευρώπη για μας, για τις μελλοντικές γενναίες οπότε πρέπει να συνεχίσεις να το κάνεις εσύ ως σκηνοθέτης. Εγώ πρέπει να συνεχίζω να το κάνω ως πολιτικός που πιστεύει στη δημιουργικότητα, στις τέχνες, ως κινητήριο δύναμη. Νομίζω λοιπόν ότι και εδώ πάλι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματος όπως και τότε που προσπαθούσαμε να αποφύγουμε το κλείσιμο του νοσοκομείου γυναικών στο Λίβερπουλ. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ανθρώπους ε, ε, σαν τον Τζέρεμι, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό που εξακολουθείς να πηγαίνει ε, σε διαδηλώσεις και να υποστηρίζει τα συνδικάτα. Πρέπει να τα κάνουμε αυτό μαζί και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό έξω από αυτό το κοινοβούλιο να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε ως Βρετανοί σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλουμε όμως εδώ να μιλήσουμε για Βρετανο, βρετανικά προβλήματα και σοσιαλιστικά προβλήματα. Δεν είναι όλα τα ίδια. Κύριε Μαλτέζε, μου έχετε ζητήσει το λόγο. Έχετε το λόγο. Κύριε Λότς, εγώ νομίζω ότι κάνατε τον ωραιότερο πολιτικό λόγο και τον πιο ε, βαθιά ευρωπαϊκό λόγο που άκουσα από τότε που εξελέγην στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ε, στην Ιταλική Αριστερά έχουμε σοβαρό πρόβλημα ηγεσία, ε, όπως και η Καθολική Εκκλησία. Αυτοί το επέλυσαν ε, εκλέγοντας λοδαπούς πάπες. Αν θέλετε να έρθετε λοιπόν να αναλάβετε τα ενία της Ιταλικής Αριστεράς, θα ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Πέρα από τα αστεία βέβαια, συμφωνώ απόλυτα με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει άρμα του νεοφιλελευθερισμού. Πρέπει πλέον να επικεντρωθούμε στα θετικά στοιχεία. Το βασικό πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι δεν είναι αρκετά δημοκρατικό. Το κοινοβούλιο το οποίο έχει εκλεγεί από το λαό έχει ελάχιστε εξουσίε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εγώ ως και εισηγητής ε, ε, για την πολιτική μου ομάδα, την ΚΟΕ, συμμετείχα στην τέταρτη δέσμη ε, μέτρων για τους σιδηροδρόμους και ο ρόλος μου ήταν να προσπαθήσω να πείσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχτεί αυτό που είχε ήδη ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει ένα κείμενο πολύ προηγμένο με πολλές εγγύσεις για τους εργαζομένους. Για παράδειγμα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες αγόραζαν ποσοστό δημοσίου σιδηροδρόμου θα έπρεπε να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για να διασφαλίσουν απασχόληση και ασφάλεια των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο τα διέγραψαν αυτά τα στοιχεία τα οποία είχε γκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η χάρτα των ευρωπαϊκών αξιών περιλαμβάνει μία έννοια που ε, δεν περιλαμβάνει αρκετά συντάγματα, την αξιοπρέπεια που είναι μία από τις πιο σημαντικές αξίες του σινεμά σας. Ε, εσείς ε, προσδώσατε εκ νέου αξιοπρέπεια σε τάξεις οι οποίες ήταν αποκλεισμένες και στις οποίες ε, αυτά τα χρόνια αυτή η πολιτική αφαίρεσε μεγάλη αξιοπρέπεια και όχι μόνο οικονομική δύναμη αλλά και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαιώματα εγγύησης. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ είναι προνόμιο για μένα να σας ακούω. Εσείς ε, παραθέσατε ε, κάτι του Μπρέκτ και εγώ θα μιλήσω για τον Μπρέκτ στο τέλος. Ε, υπήρχε μια φράση του Μπρέκτ που ανέκαθεν μου άρεσε. Λέει ότι καθόμαστε από την πλευρά του λάθους γιατί όλες οι υπόλοιπες θέσεις ήταν κατηλημένες. Και εγώ σας ευχαριστώ που εδώ και τόσα χρόνια κάθεστε από την πλευρά του λάθους. Ευχαριστώ κύριε Μαλτέζε να δώσω το λόγο στη Σελήνα, αν θέλει να πάρει το λόγο. Και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στον Κεν Λόουτς. Σελίνα, αν θέλεις. Αν θέλεις, αν θέλεις. Πες μας κάτι αισιόδοξο, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, θα πω κάτι αισιόδοξο, γι' αυτό είμαι εδώ. Θα ήθελα να πω, για να μιλήσουμε και για το βραβείο Λουξ, κάνουμε σαν ε, ο πολιτισμός, ε, η λογοτεχνία από το ένα στο άλλο κράτος μέλος πρέπει να δημιουργεί γέφυρες εμείς ε, το ξέρουμε, ε, εμείς που ταξιδεύουμε με τα έργα μας ολόκληρη στην Ευρώπη, υπάρχουν γέφυρες, είναι πάρα πολύ εύκολο να ταξιδέψει κανείς με τον κινηματογράφο, είναι σαν να ε, λέει κανείς στον κόσμο ότι πρέπει να φάνε πολιτισμό για να μπορέσουν να καταλάβουν την Ευρώπη. Όχι, αυτό το καταλαβαίνουν, τα υπόλοιπα είναι που πρέπει να τα εξηγήσουμε, αυτό είναι το δύσκολο. Οι πολιτιστικές γέφυρες υπάρχουν ήδη, το να πάει κανείς σε ταξίδι με το δικό του καινούριο έργο, εγώ σε 10-12 και νέες χώρες έχω πάει ε, χώρες έχω πάει με νέα έργα. Ε, ε, μια χαρά πηγαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε προσπάθεια να δημιουργήσουμε γέφυρες με την τέχνη. Όχι, η τέχνη είναι γέφυρα. Το θέμα είναι πώς μπορούν να κυκλοφορήσουν τα έργα. Γι' αυτό ακριβώς συζητούμε. Είναι πώς θα μπορέσουμε να κυκλοφορούν, πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αγοράς. Δεν έχουν πρόβλημα αλλιώ να κυκλοφορήσουν μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό ήθελα να πω. Επίσης, ήθελα να πω ότι προσπαθούμε να σκεφτούμε τον πολιτισμό ως παρελθόν. Είναι κάτι ζωντανό όμως, είναι κάτι σημερινό και πρέπει να είναι και πιο αντιπροσωπευτικός ο πολιτισμός ε, της σημερινής κοινωνίας. Για τις γυναίκες να πω, 80% των, ε, ε, των έργων είναι δημιουργία ανδρών, 20% ε, μόνο είναι από γυναίκες. Στη Γαλλία έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό γυναικών ε, ε, που δημιουργούν, που παράγουν έργα. Στο μικρές, μικρού μήκου ταινίε είναι όλο και περισσότερες οι γυναίκες. Θα σας πω το νούμερο αυτό γιατί εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω γιατί έχουν λιγότερα χρήματα οι γυναίκες, πολύ λιγότερα για να κάνουν μια ταινία. 2,8 εκατομμύρια για ένα έργο που το κάνει μια γυναίκα και τέσσερα αν ε, το κάνει άντρα. Και στα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ από τότε που άρχισαν ε, να υπάρχουν οι κάνες, 1.800 ε, επιλογές, 70 γυναικών. Και ναι, είναι γεγονό ότι το παρελθόν δεν υπήρχαν γυναίκες που να κάνουν ταινίες. Όμως προσφάτω έχει αυξηθεί ο αριθμό και αυτό ο λόγος ήταν ε, ότι υπήρχε συγκέντρωση εξουσίας από αυτούς που έχουν την εξουσία. Δεν ε, είναι ε, σωστό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζονται περισσότερες γυναίκες, χρειάζονται περισσότερες Άραβες, χρειάζονται περισσότεροι Άραβες, χρειάζεται περισσότερη ποικιλία, περισσότερη ποικιλομορφία για να υπάρχει μεγαλύτερος πολιτισμός. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά δεν είχαμε και πάρα πολύ χρόνο. Δεν ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάπως μας φέρνει στο δρόμο του βραβείου Λουξ, που κάνει τη δουλειά του και ως προς αυτό. Πέντε λεπτά έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας. Κύριε Λόουτς. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Λόουτς. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ διδακτική η διαδικασία και άκουσα με ενδιαφέρον όσα είπαν οι ομιλητές. Πρέπει να διορθώσω το εξή. Φοβάμαι ότι οι ταινίε δεν μπορούν να προβάλλονται δωρεάν γιατί ανήκουν στους διανομή Και εγώ αν τους δώσω μια ταινία δωρεάν, κάποιος μου το είπε αυτό, ναι. Είναι στο διαδίκτυο μεταδίδονται ζωντανά ε, δωρεάν. Αλλά εάν κάποιος πει ότι τους ανήκει τότε πρέπει να τις αφαιρέσουμε. Στη νέα ταινία όμως, ε, στη Βρετανία ελπίζουμε να προβληθεί και σε κοινότητες ε, ε, με πολύ χαμηλό Νομίζω ότι το όλο θέμα της διανομής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το πρόβλημα είναι ότι οι πρωτοβουλίες οι οποίες είναι καλοί, καλές ακόμα είναι στο περιθώριο. Στη χώρα μου αν είστε στο Λονδίνο μπορείς να δεις ευρωπαϊκές ταινίες, αν είσαι εκτός Λονδίνου σχεδόν καθόλου. Δεν συμβαίνει λοιπόν προβολή. Οι περισσότεροι δεν θα μπορέσουν να δουν τις ταινίε που συζητήσαμε. Και πιστεύω ότι αν είμαστε σοβαροί και αν θέλουμε να κάνουμε ευρωπαϊκό κινηματογράφο ο οποίος να διατίθεται σε όλους, τότε πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε ε, να υπάρχουν ε, ε, κινηματογράφοι στην ιδιοκτησία των Δήμων όπως οι Δήμοι έχουν στην ιδιοκτησία τους θέατρα και να προβάλλονται όχι από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα fast food αλλά για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τις ταινίε. Είναι πολύ σοβαρή η όλη η διαδικασία της διανομής και ξεκινά από την ιδιοκτησία του κινηματογράφου, της αίθουσας. Αυτή είναι η βασική παρατήρηση. Παρεπιπτόντω, ε, να πω ότι πολλοί λένε ότι θα ήμασταν χαμένοι χωρί τα φεστιβάλ. Αυτό το οποίο όμω είναι θλιβερό είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να διεξαχθεί φεστιβάλ πλέον χωρί να υπάρχει χορηγία από κάποια μεγάλη επιχείρηση. Και γιατί αυτό. Διότι βεβαίω καταρχά θέλουν να προβληθεί το όνομά του, αλλά η ιδεολογία που υφέρπει είναι ότι δεν συμβαίνει τίποτα χωρί τι μεγάλε επιχειρήσει. Εάν δεν μπουν το ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε καν κινηματογραφικό φεστιβάλ χωρί χορηγό κάποια πετρελαϊκή επιχείρηση επιβάλλουν την παρουσία του για να δείξουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτισμού μας. Δεν πρέπει να είναι στο επίκεντρο του πολιτισμού μας. Πρέπει να μπορούμε να διεξάγουμε φεστιβάλ, εκθέσεις, συναυλίες χωρί ε, την ε, ε, ε σύμφωνη γνώμη των μεγάλων επιχειρήσεων. Τώρα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποκλειστικά νεοφιλελεύθερη οργάνωση, ε, εγώ υποτάσαμε στις ανώτερες γνώσεις σας, εγώ κοιτάω τα γεγονότα, τις συνθήκες, τις συμφωνίες, κοιτάω τι λένε τα δικαστήρια και βλέπω τι συμβαίνει. Και πραγματικά εμένα μου φαίνεται πολύ νεοφιλελεύθερη. Μπορεί βέβαια να μην φαίνεται σε εσά από τα έδρανα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αποδείξετε ότι δεν είναι και αυτό πρέπει να γίνει με πράξεις. Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να αλλάξουν πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες και μετά να έρχεται να μου πείτε ότι δεν είναι νεοφιλελεύθεροι. Όταν συμπεριφέρεστε σε χώρες όπως η Ελλάδα με τέτοιο τρόπο, τότε πρέπει να πείτε ότι όχι, δεν πρέπει να πουλήσετε όλα τα δημόσια αγαθά σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υποχρεώνει την Ελλάδα να πουλήσει τα δημόσια αγαθά της. Αν πραγματικά θέλετε να πείτε ότι δεν είστε νεοφιλελεύθεροι, αλλάξτε τα αυτά και θα σας πιστέψω κι εγώ και θα σας πιστέψουν κι άλλοι για την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων και πάλι. Ε, η μόνη άλλη παράθεση που ήθελα να σας διαβάσω είναι μια παράθεση από τον William Blake, έναν πολύ μεγάλο ε, ποιητή, ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, ε, ζωγράφο, ο οποίος είπε Όπου υπάρχει άποψη της, ε, του χρήματος δεν μπορεί να υπάρχει τέχνη παρά μόνον πόλεμος και νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο. Uh, ναι, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους καλεσμένους μας. Ε, νομίζω ότι είσαστε πολύ αποφασιστικός ε, άνθρωπος, ε, δεσμευμένος στις υποχρεώσεις και ακόμα και αν διαφωνούμε με τις απόψεις σας, ήταν πολύ ζωντανή η συζήτηση και αυτό μας ενδιαφέρει σε ευρωπαϊκές συζητήσεις και νομίζω ότι όλοι απολαύσαμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Doris Πακ. Χαιρόμαστε που σε ξαναβλέπουμε. Και ε, να σας υπενθυμίσω συνάδελφοι και ε, στους υπολείπους βεβαίως που είναι εδώ στην αίθουσα σήμερα. Ε, σήμερα στις 7 ε, παρατέταρτο έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης 100 σκιές του φωτού για το 10η επέτειο του βραβείου Λουξ στο Παρλαμεντάριο. Ο Αντιπρόεδρος Αντώνιο Ταγιάννη και η Σίλβια Κώστα θα προεδρεύουν. Είστε όλοι καλεσμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.